Uh, Καλησπέρα σα, συναδελφοί. Και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη εμπορική διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ. Από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Και θα δώσω το λόγο στον συντάκτη τη ερώτηση, τον κύριο